θέσουμε κάποιους στόχους και ότι θα καταφέρουμε να μας δοθούν, θα μας δοθούν οι απαραίτητες δυνατότητες προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καλύτερα τους οικονομικούς μας πόρους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας με θέμα «Η κατάσταση στο Ελεφαντοστούν». Ε, Vice President, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ. αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση στην ακτή Ελεβαντοστού ε, είναι πολύ δύσκολη γιατί απειλούνται ζωέ ε, των πολιτών τη χώρα αλλά και των Ευρωπαίων που ζουν και εργάζονται στη χώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο ο ρόλο που παίζει η χώρα αυτή στην Αφρική αλλά και η πολλή δουλειά που έχει γίνει από τη διεθνή κοινότητα κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για την ενίσχυση τη επίλυση κρίσεων και την ενίσχυση τη σταθερότητας. Οι προεδρικές εκλογές αναμένονταν πολλά χρόνια. Τελικά ε, είναι προς τιμή του, των πολιτών που αποκινούμε τα Ηνωμένα Έθνη την ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και με τη βοήθεια του Προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο καταφέραμε τελικά να γίνουν αυτές οι εκλογές. Όλοι οι υποψήφοι είχαν ε, από προηγουμένως ε, αποφασίσει τους κανόνες, δηλαδή τον ειδικό αποεσταλμένο και το ρόλο του, του ε, τον κύριο Τσόι, για τη διευκόλυνση των εκλογών. Υπήρχε και μία αποστολή παρατήρησης εκλογών από, την, από τον κύριο Πρέντα, ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά του ε, και επίσης να πω ότι όντως έγιναν δημοκρατικά οι εκλογές και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα και την ομάδα του για το κουράγιο και την εξαιρετική του δουλειά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα αποτελέσματα ε, πιστοποιήθηκαν από τον ειδικό αντιπρόσωπο, από τον ειδικό αποσταλμένο, ε, αφού ανακοινώθηκαν από την εφορευτική επιστολή και ο πρόεδρος Βαρός ήταν ο πρώτος ο οποίος συνεχάρει τον Αλασάν Κατάρα για την ε, νίκη του. Η διεθνής κοινότητα τον αναγνώρισε, η ΕΚΟΒΑΣ και η Αφρικανική Ένωση ήταν ε, σαφέστατη ε, στην άποψή τους. Είναι ο νόμιμος πρόεδρος της ακτής ε, ελεφαντοστού και ε, εκείνος ήταν ε, σαφή στη δήλωσή του. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να αποδεχθούν ε, το εκλογικό αποτέλεσμα, να μην προσφύγουν στη βία, να σεβαστούν το εκλογικό αποτέλεσμα και πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, την μας στην, στην δίκαιη και δημοκρατική ανάληψη εξουσίας. Επίσης πρέπει να τιμωρηθούν όλοι όσοι παρεμποδίζουν την υλοποίηση του αποτελέσματος των εκλογών. Υπήρχαν κυρώσεις ε, για την ακτή ελεφαντοστού. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει στοχευμένα μέτρα και το έχουμε πει πολλές φορές, το είπαμε ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ότι θέλουμε να λάβουμε μέτρα για να ενισχύσουμε τις νομίμως εκλεγμένες αρχές. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται και από την κοινή γνώμη και από πολλούς εταίρους και στην Αφρική αλλά και στις γειτονικές ευρωπαϊκέ ε, χώρες, ε, οι οποίες βρίσκονται σε μια μεταπολεμική περίοδο και ε, βρίσκονται σε μια δύσκολη περίοδο εκδημοκρατισμού επειδή υπήρχε και συνταγματική κρίση στην ακτή Ελεφαντοστού και αυτό θα, αυτό θα στείλει ένα σαφέ ε, μήνυμα σε ολόκληρη την ε, Αφρικανική Ήπειρο και σε όσε χώρε είναι υπέρ και σε όσε χώρε είναι κατά του εκδημοκρατισμού. Ε, ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ω μεγάλο παίκτη, ε, η αξιοπιστία μα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι ακόμη σημαντικότερη αν μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια ειρηνική μετάβαση εξουσία με σεβασμό της απόφασης ε, των πολιτών της ακτής του Ελεφαντοστού σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές. <clears throat> Τώρα θα πάρουν το λόγο μιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Πρέντα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Euh, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία εκπρόσωπε. Ήμουνα στην ακτή Ελεφαντοστού συμμετέχοντα στην ομάδα επιτήρηση, στην αποστολή επιτήρηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα πραγματικά να χαιρετήσω το θάρρο και τη δέσμευση των παρατηρητών από 26 χώρε. Περίπου 100 άτομα, 120 παρατηρητέ που επί τόπου κάναν μια εξαιρετική, θαυμάσια δουλειά και που είδανε η διεισόμαση αυτό το οποίο έλεγαν και οι πολίτε τη ακτή του Ελεφανταστού παντού, ότι έχουμε κουραστεί πια. Αυτό λέγανε συνεχώς και ουσιαστικά μέσω αυτού ήθελαν να εκφράσουν ότι περίμεναν τι εκλογέ ω το τέλο μια πολιτική κρίση. Όλοι επιθυμούσαν η πολιτική κρίση να τερματιστεί με τι εκλογέ. Με εξαίρεση βέβαια τον απερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Γκμπάγκμπο, ο οποίο αρνήθηκε να παραχωρήσει την εξουσία και που χρησιμοποίησε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μην τελειώσει η πολιτική αυτή κρίση και ουσιαστικά με την σύμφωνη γνώμη του Συνταγματικού Συμβουλίου που είναι υπό την επιρροή του κατάφερε να κυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν υπέρ του αντιπάλου του. Και αντί να τερματιστεί τελικά η κρίση, βλέπουμε ότι η κρίση έχει γίνει ακόμα πιο πολύπλοκη. Η ισορροπία ήταν πολύ εύθραυστη και τώρα ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή μιας διένεξης. Είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρκεί να δείτε τι γίνεται με την ε, ψηφοφορία με, στα εκλογικά τμήματα και στον πρώτο και στον ε, δεύτερο γύρο και τι έγινε ακριβώς και στα στρατόπεδα. Επίσης θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την αποφασιστικότητα της ύπατης εκπροσώπου, τη δέσμευσή της υπέρ των κανόνων που θα πρέπει να ισχύουν, το ότι δεσμεύεται και το ζήτημα αυτό. Είδα ότι το Συμβούλιο είπε ότι θα υπάρχουν σύντομα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις και κάποια περιοριστικά μέτρα. Πότε ακριβώς θα εγκριθούν τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πράντα. Τώρα ε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών για τρία λεπτά η κυρία Ντοκάιζερ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο Πρεντά και την ομάδα του για την αξιοσημείωτη ε, εργασία τους και την κάθε άστον βεβαίως την ύπατη εκπρόσωπο για την αποφασιστικότητα που έδειξε μαζί με όλη τη διεθνή κοινότητα στην παρακολούθηση αυτών των εκλογών. Νομίζω ότι για όλους εμάς που θέλουμε πραγματικά να διατηρηθεί αυτό το καταπληκτικό ε, μέσω που έχουμε παρατήρηση των εκλογών υπέρ της δημοκρατίας να δίνουμε συνέχεια και χαιρόμαστε ακριβώς επειδή παρακολουθούμε τα πράγματα και δίνουμε συνέχεια σε μια προσπάθεια σφετερισμού του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό πραγματικά με ικανοποιεί πάρα πολύ και ελπίζω να ε, μεταφερθεί και σε άλλα σημεία εάν παρελπίδα φτάσουμε σε εκεί. Και τώρα θα ήθελα να πω επίσης, γιατί μου το προσάπουν πολύ όχι ο Κότρα δεν είναι ε, της Ευρώπης ο υποψήφιος. Όλη η διεθνής κοινότητα τον υποστήριξε. Η Αφρικανική Ένωση, η Οικονομική Κοινότητα της Δυτικής Αφρικής, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρώπη με μια φωνή και ε, πραγματικά και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Για τον κύριο Κόταρα τώρα ακούμε ότι βγάζει τον κόσμο του στο δρόμο. Ε, εκεί ενισχώ λίγο περισσότερο, διότι ε, δεν καταλαβαίνω ε, ποια ε, λύση μπορεί να δοθεί στους δρόμους με το σχετισμό δυνάμεων που επικρατεί. Και θα ήθελα να επανέλθω σε ένα κείμενο που είναι σε ένα στάδιο προσχεδίου στη ΣΑΚΕ και το συζητήσαμε και στην τελευταία ισομερή που είχαμε πάει μερικοί από εμά στην ΑΚΕ και είναι μια πρόκληση για το μέλλον, τη δημοκρατία και ε, για τη Διεθνή Ένωμη Τάξη. Συντάκτες είναι ένας από την κάθε πλευρά, ε, έχει μέσα πάρα πολλά ε, θεσμικά και τρεις σελίδες για το πώς θα κατανέμεται η εξουσία όταν προσπαθεί κάποιος να σφετεριστεί την εξουσία και δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Για να μην αιματοκυλιστεί η χώρα δεν λύνονται αυτά στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή βεβαίω ε, αναγνωριστεί ο νικητή των εκλογών με κάποιο τρόπο στη συνέχεια να μοιραστούν την εξουσία για να μην αιματοκυλιστεί η χώρα. Σα συνιστώ την ανάγνωση του κειμένου. Είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο και μπορεί η αφρικανική πολιτική, η κουλτούρα και ο πολιτισμός να μην ξέρει τη δημοκρατία αλλά τη διαπραγματεύσει σίγουρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων η κυρία Ντουσαρνέζ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Euh, Ευχαριστώ Μερικές ώρες μετά από την... Ε, ε γιατί έφτασαν οι υποστηρικτές του Κατάρα ε, έξω από τα γραφεία του αντιπάλου τους ε, και παρακολουθείται από την, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ηρεμία και διάλογος, αλλά αυτό, αυτό το λόγο πρέπει να τον αναλάβουν οι ηγέτες ακτής ελεφαντοστού και οι δύο υποψήφοι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρχει βιαιότητα σε μια χώρα ε, η οποία έχει υποφέρει τόσο πολύ. Δεύτερο μήνυμα. Από την αρχή η διεθνή κοινότητα, η Ευρώπη αλλά και η Αφρικανική Ένωση μίλησαν ε, με μία ενιαία φωνή και κινητοποιήθηκαν για να γίνει σεβαστό το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή η πίεση πρέπει να εξακολουθεί να ασκείται και οι κυρώσει ε, που θα προβλέπονται πρέπει να εφαρμοστούν. Ο κύριο Μπάμπο πρέπει να δεχθεί την ήττα του, αλλά ο κύριο Καταρά πρέπει να συμφιλιώσει το λαό του και να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, και να σας ζητήσω να ε, μεταφέρετε αυτό το μήνυμα. Η κυρία Ντουγόν για 1,5 λεπτό εκ μέρους των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ όπως και οι προλύσαντες συνειδητοποιώ πόσο σημαντική, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση σήμερα. Υπάρχει μια έντονη πολιτική κρίση, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο συγκρούσεων, το οποίο θα μπορούσε να λάβει χώρα και τι επόμενε ακόμα ώρε. Επομένω, προφανώ είμαι υπέρ τη ενιαία φωνή με την οποία μίλησε η διεθνή κοινότητα και Πέρα από το ότι θα πρέπει προφανώς να ισχύσει η δημοκρατία, φέρουμε και μία ευθύνη να σώσουμε τους ε, κατοίκους της Τελεφαντοστόλ, να και στείλουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ότι η Αφρική μπορεί να αλλάξει γιατί πέρα από το ζήτημα τη ασφάλεια των κατοίκων τη ακτή του ελεφαντοστού, πέρα από το ζήτημα τη μείωση των εντάσεων, που ενδεχομένω βέβαια να αυξηθεί στο μέλλον, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, και άλλε γείτονε όμορε χώρε και κατά τη διάρκεια των εκλογών και στι χώρε αυτέ, μπορεί να συμβεί το ίδιο πράγμα. Να έχουμε δηλαδή έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στου απερχόμενου προέδρου και του νέου προέδρου, του νικητέ των εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα αυτό το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και ω μήνυμα προ για άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Κονγκό, που θα προχωρήσει σε εκλογές το 2011. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της μετάβασης εξουσίας να γίνεται με τρόπο δημοκρατικό, ειρηνικό, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να Καταδικάζουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ε, παίρνουν όμοιρους, ένα ολόκληρο πληθυσμό ή οδηγούν μια χώρα σε αιματοκυλισία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση και να εξασκήσουμε την απαραίτητη πίεση προκειμένου να εκδηλωθεί η ειρήνη. Για 1,5 λεπτό Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλους μας αφορά αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ακτή ελεφαντοστού. Είναι σαφές ότι η απόφαση του Συνταγματικού ε, Συμβουλίου ε, με παραβίαση του εκλογικού νόμου για αμφισβήτηση αυτών των ε, εκλογών και το αποτελέσματο που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Φορευτική Επιτροπή καταδικάζεται από τη Διεθνική Νότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, η Κοινοβουλευτική ε, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση σε προσώπησα και Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν ε, το σεβασμό τη επίσημη τη επίσημης εξαγγελίας του εκλογικού αποτελέσματο και την ε, ανάληψη καθηκόντων ε, του νέου Προέδρου όπω τον, βάσει το αποτελέσματο που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Διαφορευτική Επιτροπή και μάλιστα επιβεβαίωσε ο ΙΕ. Όλες οι πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν σε μία δήλωσή του κοινή τη συμφωνία τους ε, επί των βασικών αυτών ε, ε, σημείων. Επίσης ζήτησαν να μην υπάρξει κλιμάτωση της βίας, για να μην υπάρξει εμφύλιος πόλεμος ενδεχομένως, κάτι το οποίο θα ήταν μια πραγματική ανθρώπινη, οικονομική και κοινωνική καταστροφή για την ακτή ελεφαντοστού, κάτι το οποίο βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί. Τώρα οι επόμενοι εγγεγραμμένοι ομιλητές. Ξεκινάμε με τον κύριο Ιακολίνο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Άστον. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αξία της δημοκρατίας, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να διαπραγματευτούμε εκλογικά αποτελέσματα. Αντιπροσωπευτικότητα, κυριαρχία, όλα αυτά αποτελούν μέτρο αξιολόγηση και αναφορά ενό δημοκρατικού συστήματο. Η δική σας εργασία αυτό ακριβώς εξολογεί, καθώς επίσης και οι ομάδες των επιτόπου παρατηρητών παρακολούθησαν μια εκλογική διαδικασία που θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει ένα οριστικό αποτέλεσμα. Η επιλογή του λαού είναι ξεκάθαρη. Και δυστυχώς βλέπουμε ακόμα ότι δεν έχει αποχωρήσει από την εξουσία ο Λοράν Γκμπάγκμπο και ότι δεν έχει πάρει τη θέση του ο Αλασάνε Ουατάρα. Αυτό είναι απαράδεκτο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι απαράδεκτο για όλους όσοι πιστεύουν πραγματικά στη δικαιοσύνη. Το ότι χρησιμοποιήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η επιρροή του Προέδρου στο Σταγματικό Συμβούλιο καταδεικνύει πραγματικά πώ έχει κατάσταση στην ακτή του ελεφαντοστού. Θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν εντάσει, αντιπαραθέσει και μια κατάσταση η οποία δεν θα είναι πλέον διαχειρίσιμη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να παραγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ζητάμε οι πολίτες οι οποίοι εκφράστηκαν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο στις εκλογές αυτές θα πρέπει να εισακουστούν, θα πρέπει οι ε, επιλογή τους να γίνει σεβαστή την εξουσία να αναλάβει ο άνθρωπος που εξέλεξαν. Η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση αυτή και ελπίζουμε ότι θα, καταφέρουμε, θα, θα ολοκληρωθεί η κρίση αυτή πολύ σύντομα και Ελπίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να στείλει το απαραίτητο μήνυμα μέσω της κυρίας Άστον με απόλυτη κυριαρχία και αποφασιστικότητα. Ο κύριος για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, Πατή εκπρόσωπο, αγαπητοί συνάδελφοι, μόλι έγιναν εκλογέ στην ακτή του η διεθνή κοινότητα ε, ανέχθηκε να αναβληθούν χρόνο με το χρόνο από το καθεστώ του Λοράν Πακμπό. Αυτέ οι επανελειμμένε αναβολέ μα είχαν ανησυχήσει και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Ελπίζουμε, ελπίζαμε όμως ότι θα επικρατήσει το δημοκρατικό πνεύμα σε μια χώρα που υπέφερε τόσο πολύ γύρω από στήρες αντιπαραθέσεις σχετικά με ε, το θέμα της ιδιότητας του πολίτη της χώρας ακτής ελεφαντοστού. Ε, έγιναν οι εκλογές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διαφάνεια και χωρίς ε, βιοπραγίες. Αυτό μας χαροποιεί και αυτό μας έκανε να ελπίσουμε ότι θα σέβονταν όλες οι πλευρές το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί υπήρξε και σεβασμός. Σήμερα δυστυχώς το δημοκρατικό αποτέλεσμα δεν το δέχεται ο ερχόμενο ε, πρόεδρο. και ε, αύριο θα πρέπει να στείλουμε μια έκκληση στον πρόεδρο ΚΠΑΚΠΟ ε, να καταλάβει ότι δεν είναι δολοπλοκία ούτε μηχανογραφία ούτε συνομοσία, απλώς η βούληση του λαού. Ενώ ζούσε στην Ευρώπη ήθελε να το θεωρούν σωτήρα της χώρας του. Οι πολίτες ε, ανέλαβαν τις ευθύνες τους και η Φορευτική Επιτροπή και ε, θα ήθελα εγώ να πω επίσης ότι και στις 3 Δεκεμβρίου στην Κινσάσα στην Ισομερή Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πήραμε μια απόφαση σύμφωνη και με τη θέση που έχουν λάβει σαφέστατα τα μέλη της Δυτικοαφρικανικής Ένωσης, Οικονομικής Κοινότητας και της Αφρικανικής Ένωσης. Το καθεστώς δεν το θέλουν ούτε πολίτες της χώρας, ούτε γείτονες, ούτε η διεθνής κοινότητα. Ε, έχει έρθει ε, η ώρα να ε, αναγνωρίσει ο κύριος Παγμπό ότι ε, εξελέγει ο κύριος Κοτά να μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα το συντομότερο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, έτσι ώστε να καταλάβει και να παραδεχτεί ο κύριος Παγμπό ότι τελείωσε το παιχνίδι. Δεν θα δεχθούμε το πείσμα του και σας ευχαριστώ. Δεν θα φτάσει στο χάος η χώρα. Ο κύριος Γκέρανς έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δεν υπήρχε το εγώ του κυρίου Κμπάμπο, θα ήταν μια πηγή έμπνευση η ακτή ελεφαντοστού για όλε τι αναπτυσσόμενε χώρε που σκοπό έχουν τη δημοκρατία. Κατά τι τελευταίε εκλογέ, ε, ο λαό τη χώρα έδειξε ιδιαίτερη πολιτική οριμότητα. Επίση, οι, διεθνεί, οργανισμοί, ε, ξεκινώντα από τον ΟΗΕ, ε, δεν εντυπωσιάζονται από τι έσχατε κινήσει ενό ανθρώπου που δεν ξέρει να χάνει. Δεν έχουν κανένα ε, άλλο τρόπο να κρατήσει την λίγη αξιοπρέπεια που ε, έχει. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λειτουργήσει σωστά σε σχέση με τη στόχευση των κυρώσεων, οι οποίες δεν πρέπει να πλήξουν το λαό, που η συμπεριφορά του ήταν υποδειγματική, αλλά τον ίδιο τον κύριο Κμπάμπο ε, και του συνεργάτες του. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Άστον τι μέτρα θα λάβουμε αν εκφυλιστεί η κατάσταση και αν η προσφυγή στη βία απειλήσει τη ζωή όλο όχι μόνο των κατοίκων της χώρας αλλά και όσων ε, ε, ε, ζουν, ξένων ζουν στην χώρα. Πώς, μπορέσουμε, πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να επιλύσουμε το πρόβλημα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρινάλντι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε εκπρόσωπε, η κατάσταση στην, ακ, ακτή του λεφαντοστού αποτελεί ένα πεδίο δοκιμών στο οποίο πραγματικά δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε μία νοθεία αυτού του μεγέθους, μία νίκη η οποία έχει κλαπεί ουσιαστικά. όχι μόνο δεν είναι αποδεκτό το να δώσουμε ούτε και ένα ευρώ από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο προς μια τέτοια κυβέρνηση η οποία δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές. Θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό η ακτή του ελεφαντοστού. Η χώρα αυτή αποτελεί πεδίο δοκιμών ακόμα και για την ε, ίδια την Αφρικανική ε, Ήπειρο και για την Αφρικανική Ένωση πιο συγκεκριμένα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το, τα, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην ακτή του ελεφαντοστού προκειμένου να ε, εμφανιστούν πάλι στην επιφάνεια κάποια στερεότυπα όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε την ακτή του λεφαντοστού για να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Οι ίδιοι κάτοικοι τη χώρας δίνουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα στον κύριο Ουτάρα για να αναλάβει την εξουσία και ένα συγγραφέας το 1998 από τη χώρα αυτή δημοσίευσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Περιμένοντας την ψήφο των αγρίων ζών». Τίτλος ο οποίος πραγματικά δείχνει ποιες ήταν οι προσδοκίες του λαού αυτού. Τώρα διαδικασία Catch the Eye. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μπασέσκου. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι εκλογέ στην ακτή Ελεφαντοστού οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι δύο υποψήφοι για τι προεδρικέ εκλογέ διεκδίκησαν και οι δύο και οι νίκη και ε, διόρισαν και πρωθυπουργό ο καθένα από αυτού. Υπάρχει μόνο ο κύριο Κουατάρα που είναι ε, ο ε, νόμιμα ε, εκλεγή πρόεδρο και θα ήθελα να ζητήσω να γίνει ζευαστό το αποτέλεσμα των εκλογών τη 20η Νοεμβρίου, ειδικότερα όταν η Εφορευτική Επιτροπή, πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ο ΟΗΕ, όλοι ε, αναγνώρισαν ε, ε, τον νόμιμο πρόεδρο. Υπήρξαν επίσης πράξεις εκφοβισμού κατά των Ευρωπαίων απεσταλμένων για την παρατήρηση των εκλογών. Η πολιτική σταθερότητα έχει ήδη σημαντικές συνέπειες. Η Αφρικανική Ένωση αποφάσισε την αναστολή της συμμετοχής της ακτή ελεφαντοστού σε όλες τις δραστηριότητες ε, του οργανισμού, ώστε να μην ε, για να μην υπάρξει και πάλι ο εμφύλιος πόλεμος το 1992. Υπάρχει λοιπόν η οδός του εκδημοκρατισμού και υπάρχει και η οδός απομόνωσης. Άλλος ή άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν φαίνεται. Οπότε, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε εσείς το λόγο να κλείσετε τη συζήτηση. Ε, thank um, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα ήδη υπόθηκαν. Ο κύριος Πρέντα μίλησε και εκείνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και την ομάδα σας για το κουράγιο και τη δουλειά σας τη διάρκεια των εκλογών αυτών και θα ήθελα πραγματικά να σας επενέσω. Δύο σύντομα σχόλια που θα ήθελα να θέσω. Βεβαίως ήρθα σε επαφή με τον ε, κύριο Μπανκιμούν ε, από την αρχή της ε, κρίσης αυτής ε, και του εξήγησα πόσο απαράδεκτη είναι η κατάσταση. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε πλήρως και Ελπίζω ε, να οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν εκεί να μην απειληθούν. Ε, έχουμε και ε, σχετικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Επίσης, ελπίζω ο κατάλογος των μέτρων να είναι έτοιμος κατά τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε να τον ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν και να διατηρήσουμε την πίεση. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος βίας και αμφιβολιών σε σχέση με το τι συνέβη. Πρέπει να είμαστε πολύ κατηγορηματικοί, πάρα πολύ σαφείς, να είμαστε όσο όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμη με τη διεθνή κοινότητα για να διατηρήσουμε την πίεση όσο το δυνατόν πιο έντονη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ε, ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Ε, κυρίες και κύριοι, έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος από αντίστοιχες πολιτικές ομάδες για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Έληξε εδώ η συζήτησή μας και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι.